εργασίες θα συνεχίσουν αύριο 10 με 1. Α, όχι, 9 με 1, 9 με 1, έκανα λάθος. Και κατόπιν μετά τις 3 το απόγευμα. Η ημερησία διάταξη θα δημοσιευθεί και στο ίντρανετ. Πέρα συνεδρίσεις, καλό σας βράδυ.